η ψηφοφορία για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευάσμων. Ε, ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. The vote. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Κόρχολα. Επόμενη είναι η έκθεση της κυρίας Ρόσπαχ όσον αφορά τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αληφτικών πόρων στη Μεσόγειο θάλασσα. Με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας και επίση εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κυρία Ρόσπαχα. Και τώρα θα έρθουμε στην έκθεση του κυρίου Γκρούτε για την υπογραφή του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της Ναγκόγια Περιευθύνης. Άρχεται ψηφοφορία υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Γκρούτε. Και τώρα θα έρθουμε στην έκθεση του κυρίου Παλώνη για τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Παλώνε. Και τώρα θα έρθουμε στην έκθεση του κυρίου Ντομένιτσι για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η πρώτη ψηφοφορία αφορά το μπλοκ 1 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται μεγάλη πλειοψηφία. Οι υπόλοιπες εννέα τροπολογίες που δεν είναι συμβατές ή δεν είναι αποδεκτές, 14 τροπολογίες που έχει υποβάλει το EFD που είναι αποδεκτές. Ωστόσο, η κυρία Sharon Bowles θέλει να πάρει το λόγο. Έχετε το λόγο, κυρία Bowles, πρόεδρος της Ah, um, σας ευχαριστώ πολύ. Οι ξεχωριστές αυτές ε, ψηφοφορίες έχουν ε, γίνει αποδεκτές ε, σύμφωνα με το περιεχόμενό τους, αλλά ουσιαστικά σπάνε την συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, η οποία έγινε στην ψηφοφορία της 17ης Δεκεμβρίου στην Επιτροπή. Μολονότι λοιπόν, άσχετα με το περιεχόμενο των τροπολογιών αυτών, θα ήθελα να σας ζητήσω να καταψηφιστούν. Ευχαριστώ. και τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Έχει γίνει έτοιμα να ψηθούν από κοινού. Δύο και έξι. Έχετε καθόλου ενστάσεις. Συμφωνεί το FED. Α, πραγματικά αυτό είναι έκπληξη. Ωραία, το ζητήσατε εσείς. Ενδιαφερόμαστε να δούμε το πώς ε, ψηφίζουν οι βουλευτές για ένα τόσο σημαντικό θέμα για το άρθρο 5. Η διαφάνεια δεν θα μας έβλαπτε. έβλαπτε. ο, ο πρόεδρος είναι υπέρ. Λοιπόν, η, τεπολογία 2 με ονομαστική ψηφοφορία έρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας απορρίπτεται 8 ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Rejected. Απορρίπτεται. We'll call the vote is open. The vote is closed. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η 33 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Θέλετε, πάρε λόγο. 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 48 άρχεται ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 49 υπέρ όχι άρχεται ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται η 50 άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 55 άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 92 άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 99 άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 105. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 109. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Rejected. Απορρίπτεται. 116. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα η πρόταση της Επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το σχέδιο νομοθετικού ψηφισματός με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Ντομένιτσι. Ο κύριος Σβόμποντα ήθελε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βρίσκω την ερμηνεία των υπηρεσιών που δεχθήκαμε πολύ περίεργη. Γιατί η κυρία Μπόλς είπε ότι αν έχουμε κάποιο συμβιβασμό και κάποιες τροπολογίες στη συνέχεια, αυτό δεν έχει απολύτως κανένα νόημα θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων πραγματικά να εξετάσει αυτή την ερμηνεία και να προβεί σε μια πιο ξεκάθαρη ερμηνεία. Γιατί αν έχουμε ένα συμβασμό δεν μπορούμε να πούμε ότι τον ε, υπερψηφίσαμε και δύο λεπτά αργότερα να τον καταψηφίζουμε. Δεν έχει, αυτό είναι παράλογο. Συμφωνήσαμε με τον Πρόεδρο ότι υπάρχει, ορισμένοι κατανοούν αυτή την υβριδική προσέγγιση. Εγώ δεν ε, συμφωνώ. Τώρα θα περάσουμε σε μια άλλη έκθεση του κ. Ντομένιτς, η οποία δεν παρουσιάζει τέτοιου είδους προβλήματα που αφορά τα, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ουσιαστικά έχουμε εδώ πέρα ακριβώς την ίδια κατάσταση που είχαμε και με την προηγούμενη ψηφοφορία. Εγώ, δεδομένου ότι συμφωνώ με την πρόεδρο Μπόλς, θεωρώ ότι ε, βρισκόμαστε ακριβώς εδώ πέρα απέναντι στην ίδια διαδικασία. Αν οι πολιτικές θέσεις δεν έχουν τροποποιηθεί, τότε οφείλουμε να προχωρήσουμε όπως ακριβώς κάναμε πριν. Επομένως, αφήνω σε εσάς διακριτική σας ευχαίρεια, κύριε Πρόεδρε, να ερμηνεύσετε την κατάσταση. Λυπούμε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να το ψηφίσουμε νομίζω ότι υπάρχει μια ανάγκη να εξεταστεί. Ωραία. Το 1 με ονομαστική ψηφοφορία, μπλοκ 1. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Το εγκρίνεται μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα θα έρθουμε στις χωριστές ε, τροπολογίες. Η τέσσερα καταρχήν. Άρχεται η ψηφοφορία. the vote? Are you all certain of your votes? As has been stated, there may be merit in some of these amendments. Όπως υπόθηκε, αυτές τις απολογίες είναι ουσιαστικές. Okay. I'm going to close the vote now. Θα κλείσω την ψηφοφορία. Είστε ικανοποιημένοι? Right. I'm Απορρίπτεται. Τροπολογία 5, μονομαστική ψηφοφορία, άρτη ψηφοφορία. Παρακαλώ. Σα. Σας ευχαριστώ. Να πω απλώς στην πολιτική μου ομάδα ότι ε, αρνητικό πρόσημο θα πρέπει να υπάρχει για τις, υπο... τροπολογίες που ακολουθούν. Μπορούμε να βεβαιώσουμε με την κυρία Μπόλ ότι έχετε την ίδια προσέγγιση στην έκθεση αυτή σε σχέση με την προηγούμενη. προσέγγιση είναι η ίδια. Τροπολογία παριθμών 5, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροποποιημένη πρόταση υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σχέδιο μαθητικό ψηφίσματος μονομαστική ψηφοφορία. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται μεγάλη πλειοψηφία. Κύριε Ντομένιτσι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς. Ήταν ιδιαίτερη η ψηφοφορία αυτή γιατί βρεθήκαμε σε μια ευαίσθητη κατάσταση. Ωστόσο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες οι οποίες υποστήριξαν αυτή τη συμφωνία και ιδιαίτερα τους κοιόδης ηγητές γιατί η συμφωνία ήταν πολύ καλή και καταφέραμε τελικά με τη συμφωνία αυτή και μετά από πάρα πολλές προσπάθειες να εγκρίνουμε το πολύ σημαντικό αυτό, την πολύ σημαντική αυτή πρόταση. Σας ευχαριστώ. And thank you for your και εγώ σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας. Πολιτέ σχέδιο για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική του κ. Βαλέσα. Το λόγο έχει ο εισηγητής Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Μετά την ψηφοφορία αυτή, το επόμενο στάδιο προτού καταλήξουμε στην ισχύ του κανονισμού τελικά, θα είναι ένας τρισμερής διάλογος με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς, επειδή υπάρχει μια σύγκρουση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα υπάρξει μια καθυστέρηση. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν ένα διοργανικό διαθεσμικό πρόβλημα που έχει να κάνει με την ερμηνεία του άρθρου 43 σημείο 3 της συνθήκης όσον αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Συμβούλιο έχει συνεχιστεί η εργασία για τα αποθέματα και έχει αρχίσει και συνεχίζει να ερμηνεύει όλες τις διατάξεις προς το δικό του συμφέρον. Θέλει το Συμβούλιο να συνεχίσει να καθορίζει τα ανώτατα όρια. Αυτό επηρεάζει τόσο την αλληλεία αλλά και τις διοργανικές σχέσεις. Επομένως θα πρέπει να καταδικάσουμε τη στάση αυτή. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. 15 τροπολογίες από κοινού από την Επιτροπή Αλίας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Βαλέσσα Περνάμε στην πληροφορία της έκθεσης του κύριου Γκάλαχερ για τη διατήρηση των ελευτικών πόρων. μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών. Ο κύριος Γκάλαχερ επιθυμεί να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος Επιτροπής Αλίας θα ήθελα να σας ζητήσω την αναβολή της ψηφοφορίας γιατί υπάρχουν ε, σημαντικά προβλήματα τα οποία φάνηκαν ε, στην ε, συνεδρίαση που έγινε χθες. Μέσω της αναβολής αυτής φαίνεται τελικά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει πολύ σημαντικές δυσκολίε όσον αφορά τα μακροχρόνια προγράμματα διατήρησης των ελευτικών πόρων. Τα προγράμματα αυτά έχουν κανονικά ω στόχο τη διατήρηση των ελευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασία. Δυστυχώ ε, για τα σημαντικά αυτά προγράμματα δεν έχει επιτευχθεί καμία σημαντική πρόοδο μετά την έναρξη, τη θέση ισχύ τη ε, συνθήκη Λισαβόνα το 2009. Και νομίζω πραγματικά ότι ε, υπάρχει μια σημαντική έλλειψη ενδιαφέροντος για το σημαντικό αυτό ζήτημα. Καθότι λοιπόν δεν έχει γίνει καμία απολύτως πρόοδος, ζητούμε από την Ιρλανδική Προεδρία να ασχοληθεί με ένα ρεαλιστικό τρόπο με το ζήτημα αυτό. Προσβλέπουμε την συνεδρίαση που θα έχουμε αύριο το πρωί με τον αρμόδιο Ιρλανδό Υπουργό και ελπίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Αλίας θα έχει επιτευχθεί μια κάποια πρόοδος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταβάλει πολύ σημαντικές προσπάθειες. Θέλουμε και εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιτευχθεί μια πρόοδος. Πρέπει επιτέλους το Συμβούλιο να σεβαστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν το είδαμε τα τελευταία χρόνια. Όσο λοιπόν δεν έχει εγκριθεί ο κανονισμός αυτός, ο βασικός κανονισμός του 1998 θα συνεχίσει να ισχύει. Δυστυχώς η Ιρλανδική Προεδρία δεν έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να χαρτογραφήσει του πώς ακριβώς θα σημειωθεί πρόοδο στο μέλλον. Επομένως, εμείς δεν έχουμε καμία άλλη εναλλακτική από το να μπλοκάρουμε αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε άλλη νομοθετική διαδικασία. Εν κατακλείδη, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι ενδεχομένω ανάλογα έτοιμο να κάνω και το Φεβρουάριο, αν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα δεν επιτευχθεί πρόοδο. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση όμω να προκαταβάλω τώρα τι συζητήσει που θα γίνουν με την Προεδρία. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να ζητήσω ονομαστική ψηφοφορία για το ζήτημα αυτό τη αναβολή τη έγκριση εκθεσή μου. Σα ευχαριστώ. Χρειαζόμαστε ένα ομιλητή υπέρ τη πρόταση αναβολή τη πλειοψηφία. Υπάρχει κανείς που θέλει να μιλήσει υπέρ της αναβολής. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ στηρίζω το όσα είπε ο εισηγητής. Αυτό θα εξασφαλίσει μια ουσιαστική αναθεώρηση της ε, αλληλευτικής πολιτικής, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανακάμψουν τα αλληλευτικά αποθέματα και να έχουμε καλά διαχειριστικά σχέδια για την αλληλεία μελλοντικά. Θέλει κάποιος να μιλήσει κατά της πρότασης αναβολής. Δεν υπάρχουν εθελοντές, άρα λοιπόν θα υποβληθεί σε ψηφοφορία, νομαστική ψηφοφορία. Πρόταση να αναβληθεί η ψηφοφορία. And τη ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ε, συγχαρητήρια κύριε Γκάλαχερ με 679-677. Καλή επιτυχία σε διαπραγματεύσει. Το επόμενο είναι η έκθεση του κυρίου Καζίνη για την τροποποίηση του κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την τάξη των αντιπροέδρων που εκλέγονται διαβοή. Θα ψηφίσουμε το κείμενο. Χρειαζόμαστε μια ειδική ε, πλειοψηφία. Ε, η τροπολογία 2 υπέρ παρακαλώ. Κατά θα ελέγξουμε, θα επαληθεύσουμε. Η ε, τροπολογία υπερθμών 2. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Νομίζω ότι απορρίφθηκε παρόλα αυτά. Γίνεται έλεγχος. Uh, Απορρίφθηκε με 492 ψήφους. Η τροπολογία 2 έχει απορριφθεί. Έχουμε την 4, την 5 και την 8. Κύριε Καζίνη, θέλετε να πάρετε το λόγο. Η τροπολογία υπαριθμών 3. Παρακαλώ κύριε Καζίνη. Κοιτάξτε, ήδη είπα ότι απορρίπτουμε το 2, 3, 4 και 5. Για το 6 είμαστε υπέρ του αρχικού κειμένου της Επιτροπής και είμαστε υπέρ του 1. Είμαστε κατά τον άλλον απλό. Well, it's not that simple, but anyway. Ε, δεν είναι και τόσο απλό, εν πάση περιπτώσει. Κάποιοι γνωρίζουν ότι θα χάσουν τις ψηφοφορίες αυτές. Οι τρία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τέσσερα και πέντε έχουν καταπέσει μάλλον. Περνάμε τώρα στην έξι. Ποιοι είναι υπέρ της έξι παρακαλώ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το 8 έχει καταπέσει θέτω σε ψηφοφορία τώρα την πρόταση απόφασης με απλή πλειοψηφία ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή Τώρα περνάμε στην έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης για την εγγύηση ε, για τους ε, νέους. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Πέντε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 2, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Παράγραφος 2. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. Τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4 σε 2 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Παράγραφος 5 σε 2 τμήματα. Πρώτο τμήμα της 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Τροπολογία 8, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος στην τροπολογία 8, ψηφίζεται. Πέραστη στις ψηφοφορίες. Απερίφθη. Τροπολογία 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέτω σε ψηφοφορία τώρα την πρόταση ψηφίσματος. Ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Πέρα τη ψηφοφορία. Δίκτυ ευχαριστώ επίσης και τις ε, αρμόδιες επιτροπές. Περνάω στην έκθεση Κολάσκα Μπομπίνσκα για το ρόλο της πολιτικής συνοχής και τον τομέα της ενέργειας. Η κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα έχει ζητήσει το λόγο. Ήταν μια ερώτηση χωρίς ε, μικρόφωνο, δεν την ακούσαμε. Θα ήθελα να πάρω το λόγο εφόσον γίνει δεκτή έκθεσή μου, λέει η κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα. Λοιπόν, ονομαστική ψηφοφορία για το 5, την τροπολογία 5 ψηφίζεται. Πέρα ψηφοφορία. Απερίφθη. Τροπολογία 1, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζεται. Πέρα ψηφοφορία. Απερίφθη. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία ονομαστική. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Έρχομαι τώρα στην παράγραφο 3, σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Το δεύτερο τμήμα της 3, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Το τρίτο τμήμα της 3 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Παράγραφος 6 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 14 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, α, Ονομαστική ψηφοφορία λοιπόν για το πρώτο τμήμα. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. Ονομαστική και για το δεύτερο τμήμα της 14 ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Παράγραφος 25. Σε δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτό. Το δεύτερο τμήμα 25 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Παράγραφος 26 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Παράγραφος 32 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Παράγραφος 35 υπέρ κατά αποχές δεν ήταν ξεκάθαρο. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 35. Ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. 37 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 42 υπέρ. Α. Ονομαστική ψηφοφορία διορθώνει ο πρόεδρος για την 42. Πέρασης ψηφοφορίας. Απερίφθη. Περνάω τώρα στη 43 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Από... Α. Ξαναρχίζω λέει ο πρόεδρος. 43 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Παράγραφο 46. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απερίφθη. 48 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 2 λοιπόν. Ψηφίζουμε. Απερίφθη. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Θέτω σε ψηφοφορία το H λατινικό σε ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα του H ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Το δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Περνάμε τώρα στο σύνολο του ψηφίσματος ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζεται. Πέρα της Τώρα, κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα, υπάρχει πλειοψηφία. Έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, τη Δευτέρα το ελεγκτικό συνέδριο ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα στον τομέα της αποδοτικότητας της ενέργειας για την ενέργεια σε ορισμένες χώρες. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει την, την έκθεση αυτή και τις συστάσεις μου υπόψη όταν προετοιμάζει την επόμενη προγραμματική περίοδο. Δεν θέλουμε εμείς τα χρήματα της συνοχής για την ενέργεια να πηγαίνουν χαμένα. Σας ευχαριστώ. Okay. Well, thank you Ευχαριστώ για το σχόλιο σας. Οι συνάδελφοι το τα άκουσαν. Τώρα η Επιτροπή φαίνεται απασχολημένη, αλλά θα διαβάσει την αποτελέσματα της ψηφοφορίας όταν τους τα στείλουμε. The next item is the vote on the report by Mrs. Goulard. Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση της κυρίας Γκουλάρ. Τροπολογία 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Πέραση της Δεκτό. Όλα τα άλλα καταπίπτουν συνεπώς. Τελειώσαμε τις ψηφοφορίες. Καλή σας όρεξη και καλή χρονιά. Uh, Συνεχίζουμε αμέσω. Επεξηγήσει ψήφου. Πρώτο για το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων των Ολομπελιών. Κύριε Σόντεγκαρτ.